Ladies Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάμε τώρα στο σημείο 17 της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Τη συζήτηση για το σημείο αυτό διοργανώνουμε μαζί με του φίλου από την Υποεπιτροπή για την Ασφάλεια και Άμυνα και σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία για τι σχέσει με την Κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ την κυρία Λουαζό, την ε, πρόεδρο τη Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ, κάθε δίπλα μου. Ένα θερμό καλωσόρισμα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Γιάνν Στόλτεμπερκ, Γενική Γραμματεύ Καλώς ήρθατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας είχαμε ξαναδεί ως προσκεκλημένο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην της νέας αστητείας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ε, προσέλευσή σα μετά την ε, ανάληψη καθηκόντων του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο για να συζητήσουμε για τα θέματα ασφάλεια και άμυνα. Στι εισαγωγικέ μου παρατηρήσει θα παραμείνω πολύ σύντομο. Απλώ να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή Εξωτερικών Προθέσεων, καθώ και η Επιτροπή Άμυνα και Ασφάλεια έχουν εργαστεί εντατικά για να εντοπίσουν ε, σημεία ε, εγκύτερης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ξέρουμε ότι η ασφάλεια και η άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ και την διατλαντική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά. Έχετε το λόγο κύριε Γενική Γραμματέα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ David και ευχαριστώ πολύ και τους προέδρους των ε, επιτροπών λοιπόν ΑΦΕΤ, ε, ΣΕΝΤΕ και της Ευρωεπιτροπής για τις αντιπροσωπείες για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ε, βλέπω πολλά νέα πρόσωπα, βλέπω όμως και κάποια οικεία από την περασμένη φορά που είχα έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ για διαφορετικού λόγου. Πρώτα απ' όλα αισθάνομαι ότι είμαι σπίτι μου. Αισθάνομαι άνετα μεταξύ βουλευτών. Υπήρξα και εγώ ίδιο βουλευτή επί 20 χρόνια και πραγματικά αυτό το σύμβολο και η έκφραση τη δημοκρατία μου αρέσει. Διότι ξέρουμε ότι οι βουλευτέ παραδοσιακά έχουν διαφορετικέ απόψει για διαφορετικά ζητήματα και παρόλα αυτά πιστεύουμε όλοι στα θεσμικά όργανα. Τη Βουλή, το Κοινοβούλιο, την έκφραση, τη δημοκρατική έκφραση ενό λαού. Τα κοινοβούλια είναι σημαντικά για όλα τα έθνη μα στι διάφορε χώρε, αλλά για και σαφώς είναι ε, εξίσου σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο για να διαμορφωθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Για σας που είστε οι βασικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Ε, και εδώ βεβαίως πρέπει να περάσω και στο επόμενο σημείο. Εγώ είμαι υπέρμαχος της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Ε, Νομίζω ότι ακόμα απομένουν πολλά σημαντικά να κάνουμε και νομίζω ότι ε, έχω πολύ καλέ σχέσει με την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ούρσουλα Φοντερλά είναι Υπουργό Άμυνα, ήταν στενή συνεργάτη σε πολλά χρόνια. Ε, και ο κύριο Μισελ. Και την περασμένη εβδομάδα συνάντησα του Υπουργού Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Τον είπα το εκπρόσωπο Μπορέλ. Και σε δύο-τρει εβδομάδε ο Γιωσέφ Μπορέλ θα έρθει στην Υπουργική Σύνοδο Υπουργών Άμυνα του ΝΑΤΟ. Οπότε συναντιόμαστε σε διαφορετικού σχηματισμού και επίπεδα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δείχνει πόσο στενή συνεργασία υπάρχει μεταξύ ημών και ημών. Είμαστε δύο διαφορετικοί οργανισμοί βεβαίω. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τις διαφορές μας, τη διαφορετικότητά μας ε, και τι αποφάσει που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Καλωσορίζω όμω το γεγονό ότι παρά τι διαφορέ μα μπορούμε να παραδεχτούμε ότι είναι εξαιρετική σημασία να στεκόμαστε ο ένα δίπλα στον άλλον, να πορευόμαστε μαζί και από πέρσι ανεβάσαμε σε επίπεδα ανίποτη ένταση τη συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ ε, τουλάχιστον περισσότερο από ό,τι ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονό ότι είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε για θέσει όπω η κυβερνοασφάλεια, οι υβριδικέ απειλέ, ότι έχουμε ασχοληθεί πολλά χρόνια μαζί με τα Δυτικά Βαλκάνια, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Αυτά δείχνουν τη σημασία που έχουν ε, τα σχετικά θέματα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τον ΝΑΤΟ. Καλωσορίζω το γεγονός ότι λόγου χάρη Έχουμε έξι σκάφη που βοηθούν να εφαρμοστεί η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση των μεταναστών. Στην Μεσόγειο έχουμε την επιχείρηση Σοφία και βεβαίως μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα για να παράσχουμε περισσότερη στήριξη εφόσον χρειαστεί αυτό για να μπορέσουμε λόγω χάρη να κοιτάξουμε κατά πόσο τηρείται το εμπάργκο των όπλων προ τη Λιβύη. Υπάρχουν διαφορετικέ λοιπόν επιχειρήσει και προσπάθειε που κάνουμε μαζί. Είναι πολλέ οι περιπτώσει που συνεργαζόμαστε. Είναι γεγονό λοιπόν. Ναι, είμαστε δύο διαφορετικοί οργανισμοί μεν. Όμω εργαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο μαζί, στενά, δε. Ε, πρέπει να ξεκινήσω λοιπόν λέγοντα ε, και επενώντα την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ΝΑΤΟ που μπόρεσαν να οργανώσουν περισσότερες κοινέ δραστηριότητες, κοινέ επιχειρήσεις. Αυτά απεικονίζουν τη σημασία της συνολική μας συνεργασίας. Η συνεργασία μας αυτή πραγματικά είναι κάτι στο οποίο πιστεύω βαθιά, γιατί πιστεύω και στη συνεργασία Βόρειας Αμερικής Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται στενά μεν, από την άλλη πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι και η Ευρώπη με τη Βόρεια Αμερική συνεργάζονται στενά δε. Πιστεύω στον διατλαντικό δεσμό, στη σχέση Ευρώπης-Βόρειας Αμερικής παρά το γεγονός ότι κάποιοι αμφισβητούν την δύναμη και την ε, ε σοβαρότητα της σχέσης αυτής. Η διατλαντική αυτή σχέση ε, νομίζω ότι ενσαρκώνεται από το ίδιο το ΝΑΤΟ, όχι μόνο την διατλαντική σχέση Βορείας Αμερικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας διατλαντικός οργανισμός και αυτή η διατλαντική σχέση, αυτός ο δεσμός ισχύει παρά τις διαφορές μας και τις διαφωνίες που βλέπουμε σήμερα να προκύπτουν. Υπάρχουν διαστάσεις απόψεων, υπάρχουν διαφορές μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης για θέματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, όπως τα εμπορικά, όπως η Πυρηνική Συμφωνία των Πυρηνικών ε, και πολλά άλλα. Ε, υπάρχουν ε, διαφορές σε διαφορετικά ζητήματα. Όμως τη διατλαντική συνεργασία την πιστεύουμε παρά τις διαφορές αυτές και πρέπει να βαδίζουμε χέρι-χέρι, διότι είμαστε ασφαλέστεροι, προστατευμένοι όταν μπορούμε να κινούμαστε μαζί και να αντιμετωπίζουμε από κοινού κοινέ απειλές διότι το περιβάλλον διαρκώ μεταβάλλεται και η συγκυρία είναι σημαντική. Έχουμε λοιπόν κοινά συμφέροντα ως σύμμαχοι, ε, συμφέροντα που αφορούν την ειρήνη και την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε και όχι να αποδυναμώσουμε τον διατλαντικό αυτό δεσμό που μας ενώνει. Ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμω και κάτι το παράδοξο, παρά τι διαστάσει απόψεων. Και κάποιοι από εσά θα έχετε ερωτήσεις, φαντάζομαι, στη συνέχεια στις ερωτήσεις σας για τις διαφορές αυτές σε διαφορετικά θέματα. Παρά τις διαφορές αυτές. Υπάρχει ένα παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι ε, τις διαφορές μας τις γεφυρώνει μια συνεργασία που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ κάνουν αυτό το που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, μάλιστα, ενώ αυτή η εντύπωση δίδεται, δεν ε, παρασύρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. σα ίσα, ο ψυχρό πόλεμο μειώθηκε και τα επίπεδα ένταση έπεσαν χάρη ε, στον περιορισμό τη παρουσία στην Ευρώπη. Δεν έχει λοιπόν ε, μειωθεί η παρουσία, αλλά έχει αυξηθεί η παρουσία των στην Ευρώπη. Με περισσότερα στρατεύματα, με περισσότερο εξοπλισμό, με εδώ και κάποιες εβδομάδες μεγάλες ασκήσεις, κοινέ ασκήσεις. Το Europe Defender 2020. Ε, Σε αυτή την άσκηση, η ΕΠΑ θα εκδιπλώσουν 20.000 ε, άνδρες, ε, στρατεύματα απευθείας από τις ΕΠΑ στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη στρατευματών από το τέλος του ψυχρού πολέμου. Άρα και πάλι είτε σας αρέσει είτε όχι, είτε είστε υπέρ είτε κατά, είναι λάθος στοιχείο να λέμε ότι είπα έχουν λιγότερη σχέση με την Ευρώπη. Έχουν περισσότερα στατεύματα τώρα στην Ευρώπη από ό,τι ποτέ στο παρελθόν. Οπότε οι ΙΠΑ δεν απομακρύνονται, πλησιάζουν, δεν μειώνουν, αυξάνουν. Και οι Ευρωπαίοι αυξάνουν την ένταση του συσχετισμού μας. Νέες δυνάμεις, νέα στατεύματα ε, στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, επίταση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μετά τις περικοπές του αμυντικό εξοπλισμού μετά τον ψυχρό πόλεμο, από όλου του συμμάχου του ΝΑΤΟ άλλωστε, τώρα όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αρχίζουν να, αυξάνουν, να αυξάνουν τον αμυντικό του εξοπλισμό. Δεν λέω ότι έχουν επενδύσει όσα θα έπρεπε. Λέω όμω ότι η διαφορά είναι μεγάλη. Από τη μείωση που είχαμε πριν πάμε σε αύξηση. Και είναι γεγονό ότι όλοι οι σύμμαχοι, όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδά επενδύουν περισσότερα στην άμυνα. Από το 2016 μόλις η Ευρωπαϊκή Συμμαχοί έχουν προσθέσει 130 δις, 130 δις αμερικανικά δολάρια περισσότερα για την άμυνα. Σοβαρότατη αύξηση. Εάν δείτε μάλιστα τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο το Δεκέμβριο και το τι υπόθηκε εκεί, το μήνυμα που προέκυψε και από τη ΣΥΠΑ ήταν, ήταν ότι αναγνωρίζουν αυτή την πρόοδο και τονίζουν ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι οι επενδύσει γίνονται στον ευρωπαϊκό ε, εξοπλισμό και τον ευρωπαϊκό αμυντικό εξοπλισμό. Όχι για να ικανοποιήσουν την Αμερική, την συμμαχία. Είναι προ ε, όφελο των Ευρωπαίων να το πράξουν αυτό. Και μάλιστα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αποφάσισαν ε, ήδη από την Σύνοδο του Λονδίνου το 2014 να αυξηθεί ο αμυντικός εξοπλισμός και οι επενδύσεις εκεί. Παρά λοιπόν τα ερωτηματικά που υπάρχουν για το κατά πόσο ο διατλαντικός δεσμός είναι ισχυρός ή όχι, είναι άρρηκτος, έχει ενισχυθεί και όλα τα τελευταία χρόνια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε περισσότερα μαζί από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Καλωσορίζω το γεγονός αυτό και Χρειαζόμαστε ε, την Βόρεια Αμερική μαζί με την Ευρώπη να συνεργάζονται ε, στο επίπεδο του ΝΑΤΟ για τον διατλαντικό αυτό δεσμό, αλλά θα τις χρειαστούμε και στο μέλλον μαζί για να αντιμετωπίζουμε και παλιές και νέες προκλήσεις. Πολύ σύντομα να αναφέρω μερικές. Πρώτον, καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα και πολλοί λόγοι να ανησυχούμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η συνεργασία Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης έχουν επιτρέψει να γίνουν πολλά βήματα πρόοδου. Ε, πριν από λίγους μήνες ε, το ISIS ε, ήλεγχε μια επικράτεια που ήταν μεγάλη στον Αμένο Βασίλειο με εκατομμύρια κόσμο και βλέπαμε τη βαναυσότητα αυτού του οργανισμού. Αποκεφάλιζαν κόσμο, ο βιασμός ήταν στρατιωτικό όπλο, η δουλεία, η σκλαβιά βαναυσότητα που ξεπερνούσε κάθε όριο της φαντασίας. Τώρα ε, υπάρχουν ολόκληρε περιοχέ που έχουν απελευθερωθεί. Το ΑΕΖΙΣ έχει χάσει τον έλεγχο των περισσότερων εδαφών και του κόσμου που μέχρι τώρα είχε υπό την ε, ε, κατοχή του. Αυτό χάρη στι κοινέ προσπάθειες βόρεια Αμερική και Ευρώπης, που είμαστε σύμμαχοι. Δεν είναι κάτι μικρό αυτό, είναι τεράστιο. Απέτησε τεράστιες προσπάθειες. Απλώς να σας πω ότι μου φαίνεται ότι κάπως μας διαφεύγει τι μεγάλο κίνδυνο χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Ιράκ όμω, γιατί η καταπολέμηση και η μάχη κατά του Άιζες δεν έχει τελειώσει. Είμαστε μια παγκόσμια συμμαχία λοιπόν μπορεί να νικήσει και νίκησε σε ένα βαθμό το ΝΤΑΕΣ. Ε, και ε, έχουν πάυσει οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προς το Ιράκ. Έχουν ανασταλεί, αλλά πρέπει να ξαναρχίσουν ως τα δυνατόν συντομότερα, διότι το Ιράκ χρειάζεται στήριξη. Θα πέσει πάλι σε παγίδα ένοπλη σύγκρουση ε, το Ιράκ, εάν δεν βοηθήσουμε και μπορεί να επιστρέψει το Άιζης. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Και είναι πολλά αυτά που θα μπορούσα να πω. Απλώ να μοιραστώ μαζί σα μία σημαντική σκέψη, ένα μήνυμα όταν κοιτάζω τι περισσότερο μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ, η Δύση, αυτή η διεθνής, ε, η παγκόσμια συμμαχία που είμαστε εμεί, πρέπει να στραφούμε ε, στο κατά πόσο μπορούμε να έχουμε περισσότερε πολεμικέ επιχείρησει. Διότι ε, το ΝΑΤΟ πρέπει να μπορεί να ασχολείται και να οργανώνει πολεμικέ επιχειρήσει από όσο χρειαστεί. Στα Βαλκάνια, στο Ιράκ και το καθεξή. Όμω. καλύτερο θα ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα στι τοπικέ δυνάμει, να αναλάβουν δράση κατά των τρομοκρατών οι ίδιοι, να ε, δράσουν τοπικές ε, δυνάμει. Πάντοτε δρούμε ως εξωτερικοί παρεμβαίνοντε. Το βασικό λοιπόν που μα απασχολεί στο ΝΑΤΟ δεν είναι απλώ να διοργανώνουμε μεγάλε πολεμικέ επιχειρήσει, αλλά να εκπαιδεύσουμε και να οικοδομήσουμε τοπικέ δυνατότητε όπω κάναμε στο Αφγανιστάν, όπω κάνουμε στο Ιράκ και όπω και πάλι θέλουμε να κάνουμε με άλλους συμμάχους ε, στην περιοχή, την Ιορδανία, την Τινησία να έχουν δυνατότητε, ειδικέ δυνατότητε και μυστικέ υπηρεσίε για να μπορούν να καταπολεμήσουν του τρομοκράτε. Η πρόληψη είναι καλύτερη από την παρέμβαση, λέμε. Το να οικοδομήσουν ίδιε δυνατότητε είναι καλύτερο από το να πηγαίνουμε μετά για να θεραπεύουμε ένα πρόβλημα. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να διαδραματίσει, είναι παρούσα και πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει όχι μόνη της, μαζί με τη Βόρεια Αμερική. Το δεύτερο στοιχείο, η δεύτερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού είναι η Ρωσία. όπως θα ξέρετε στο ΝΑΤΟ έχουμε την ε, προσέγγιση διπλής ταχύτητας ε, προς τη Ρωσία. Πρώτα απ' όλα την άμυνά μα και δεύτερον το διάλογο. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, συσπηρωμένοι, δυνατοί και να μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα και με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι δυνατή και θα μείνει παρούσα και δυνατή για πολύ καιρό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε επικοδομητική σχέση μαζί του ο διάλογο. Δεν είναι δείγμα δυναμία, είναι δείγμα δύναμη. Και βεβαίω χρειαζόμαστε και τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά από κοντά. Ε, πρέπει η Βόρεια Αμερική να βοηθήσει για να είμαστε αξιόπιστοι εταίροι και στα θέματα άμυνα. Όμω χρειαζόμαστε τη Βόρεια Αμερική οπωσδήποτε για να είναι ε, ε, ουσιαστικό ο διάλογο μα με τη Ρωσία. Ιδάλω, ένα μεγάλο τμήμα του διαλόγου αυτού για τον έλεγχο των όπλων δεν έχει νόημα. Ο έλεγχο των όπλων πρέπει να έχει ε, γύρω από το τραπέζι τη συζήτηση και τη είπα. Δηλαδή, η, η απομάκρυνση από τη συνθήκη για την χρήση των πυρηνικών όπλων και την εξάπλωση των ε, μακραίους βεληνικούς, μεγάλου στην Ευρώπη είναι μια συμφωνία που ξεκίνησε από ΕΠΑ και Ρωσία. Αλλά έχει κάθε λόγο ύπαρξη για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ουσιαστικός ε, έλεγχος των όπλων και σίγουρα πρέπει να είναι παρούσε οι Ηνωμένε Πολιτείες προχωρώ, διότι από ό,τι βλέπω πρέπει να αφήσω χρόνο και για ερωταπαντήσεις. Τρίτη πρόκληση που θα αναφέρω ε, εντάχει είναι μια νέα, οι νέε αναδυόμενες μάλλον απειλές συνολικά. Τεχνολογικές, από την τεχνητή ευφυΐα, οι αυτόνομες πλατφόρμες όπλων, τα μεγάλα δεδομένα, big data, όλες αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογικές λύσεις θα αλλάξουν την φύση των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως και η βιομηχανική επανάσταση στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε όλοι μας την επινοητικότητα ε, και την ε, δημιουργικότητα για να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή παρακολούθησης αυτών των εξελίξεων και να είμαστε τεχνολογικά προετοιμασμένοι. Αυτό συνδέεται και με την ε, περίπτωση της αντιδιαστολής Ρωσίας-Κίνας. Είναι στην αιχμή των εξελίξεων η χώρα αυτή. Η τεχνητή ευθεία στην Κίνα είναι πολύ προηγμένη ε, και με μεγάλες επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμαστε και στα θέματα αυτά και να κοιτάζουμε την ε, άνοδο της Κίνας εκεί. Υπάρχουν ευκαιρίες αλλά και σοβαρά προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Κίνα έχει το, δευτερο, μεγαλύτερο αμυντικό εξοπλισμό στον κόσμο. Τα τελευταία πέντε χρόνια είχαν 80 νέα πολεμικά σκάφη. Ε, το σύνολο των Βρετανικών σκαφών, του πολεμικού στόλου της Βρετανίας. Μόνο σε πέντε χρόνια το κάνανε αυτό οι Κινέζοι. Φανταστείτε. Ε, κάποιοι και στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική λένε πόσο μεγάλο η Κίνα. Έχει ανασυχητικό μέγεθος. Πρέπει γι' αυτό λοιπόν να σταθούμε μαζί Βόρεια Αμερική και Ευρώπη. Το 50% του ΑΕΠ και των αμυντικών εξοπλισμών μπορούμε να το καλύψουμε εμείς. Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική είμαστε οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφωνίες, όμως εφόσον σταθούμε ο ένας στο πλευρό του άλλου και μπορούμε την κοινή μας ασφάλεια, την κοινή μας προστασία να τα αντιμετωπίσουμε από κοινού, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Μπορεί να είναι ισχυρό ο διατλαντικός δεσμός και μπορούμε να έχουμε και ένα δυνατό, ένα ισχυρό ΝΑΤΟ για να έχουμε και μια αποτελεσματική ενεργή συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης εγώ Αμερικής και ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Excellent. Thank you, Secretary General. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενική Γραμματέα. Έχουμε τώρα περίπου 35 λεπτά στην ε, διάθεσή μας για μια ανταλλαγή απόψεων. Έχω έναν μακροσκελέστατο κατάλογο ομιλητών, πάνω από 30 μέλη ε, θα πάρουν το λόγο. Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους όσοι θα το ήθελαν θα δώσω προτεραιότητα στου συντονιστέ, ζητώ την κατανόησή σα, Πρώτον, θα δώσω το λόγο στον ε, πρόεδρο της αντιπροσωπείας μας για τις σχέσει ε, με την Νατοική Κοινοβουλευτική ε, Ολομέλεια, με τον, στον κύριο Πέτρες. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Στόλτεμπεργκ που είστε εδώ σήμερα και μας δίνετε όλες αυτές τις πληροφορίες. Δύο σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, διάβασα το πρόεδρο Τραμπ θέλει να επεκταθεί το ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. Ποια είναι η δική σας ε, γνώμη σε σχέση με αυτή την πρόταση. Δεύτερον, ως πρόεδρος ε, της ε, αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στο ΝΑΤΟ, ξέρετε ότι έχουμε μία θέση ζωή Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου όπως άλλοι πρόσωποι εθνικών κοινοβουλίων. Μήπως έχει έρθει η ώρα να αναβαθμιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αντιπροσωπεία του. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Πολύ καλά ερωτήματα, Κρίς. Ευχαριστούμε και έδωσε και το καλό παράδειγμα σε ό,τι φορά το χρόνο. Αν συμφωνείτε, καλό είναι να κάνουμε ένα γύρο ε, των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Γκάλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, εν γέννη συμμεριζόμαστε ε, την ανάλυση της σημερινής κατάστασης που κάνατε. Σε μία από τις προηγούμενες παρεμβάσεις εδώ είχατε πει ότι υπάρχουν ε, τομείς συνεργασίας, ανθεκτικότητα μεταξύ ημών, ανθεκτικότητα με τους ε, γείτονες και ενίσχυση των συνόρων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δεν έχουμε δράσει ο ένα απέναντι στον άλλον σε ό,τι αφορά την ε, θέσπιση του Ταμείου Άμυνα. Ε, θεωρείτε ότι έχει πάει καλά αυτή η συνεργασία. Μετά γνωρίζετε ότι η στρατηγική αυτονομία είναι ένα όρο ε, που δημιουργεί αναστάτωση στους νατοικούς κύκλους κάποιες φορές. Συμφωνείτε ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε από μόνοι μας, επειδή αναφερθήκατε στη Λιβύη, αλλά και η Τουρκία μπορεί να μην ακολουθεί 100% τη δική μας γραμμή. Τι θα κάνουμε αν δεν έχουμε δυνατότητα να καταφύγουμε σε ανατοϊκού πόρου αν η Τουρκία πει όχι. Θεωρείτε ότι αυτό από μόνο του απαιτεί στρατηγική αυτονομία, προκειμένου και εμεί να μπορούμε να κάνουμε στη Λιβύη αυτό που πρέπει. Ευχαριστούμε από του σοσιαλιστές ο Τονίνο Πίτσουλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, καλώ ήλθατε και πάλι στο Κοινοβούλιο, όπως πάντα, είναι δύσκολη καιρή που περνούμε και είναι σημαντικό να διατηρήσουμε συνοχή και ενότητα στα μέλη του ΝΑΤΟ. Επειδή γνωρίζουμε και τις τουρκικές ενέργειες στη Βόρεια Συρία, τις ε, διαδικασίες που ακολουθεί η Τουρκία και οι ενέργειές της στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά που δεν συνάδουν ε, με την ε, νατοική πολιτική συνοχή. Εσείς πώς βλέπετε ε, τον ρόλο της Τουρκίας σήμερα, καθότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, πώς βλέπετε τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία και εφόσον βλέπουμε ότι αυξάνεται η επιρροή στην περιοχή και ότι η Τουρκία πρόσφατα αγόρασε και ένα σύστημα αντιπυραυλικό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κιουτσούκ από την ομάδα Ρενιού. Α, Πέτρας, συγγνώμη. Ευχαριστώ, David. Κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας. Η ομάδα μας ε, προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασία μαζί σας ε, στις γραμμές που αναφέρατε. Εμείς είμαστε υπέρ των περαιτέρω εξελίξεων για την ε, Ένωση Άμυνας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα 22 μέλη που είναι κοινά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ε, θα σταθούν από κοινού λοιπόν ε, εν ώψη των μελλοντικών προκλήσεων. Θα ήθελα να σχολιάσετε ε, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, δυστυχώς. Ποια είναι η δική σα θέση, τι θα μπορούσε να γίνει, προκειμένου να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ως ασθενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλήρες μέλος βεβαίως του ΝΑΤΟ. Κατά τη δική μου γνώμη υπάρχει τώρα μια πρόκληση όχι μόνο σε σχέση με τις ευρωατλαντικές ε, σχέσεις μόνο αλλά και μεταξύ των δύο ε, όχθων της ε, μάχης. Μετά ένα σχόλιο για τους ε, ομοειδεάτες ε, εταίρους μας που μπορούμε να καλέσουμε σε όλες τις ενέργειες και δραστηριότητές μας που είναι απαραίτητες ε, ανά τον κόσμο για την επίτευξη της ειρήνης και σταθερότητας. Ποιος είναι αυτός ο κατάλογος. Ελπίζω να είναι μεγάλος. Ευχαριστούμε Πέτρας. Πιατικόβα για τους πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα που είστε εδώ σήμερα μαζί μας τρία ερωτήματα εντάχει. Το ΝΑΤΟ πρόσφατα για πρώτη φορά έδειξε το ζήτημα της Κίνας. Εδώ κάθομαι. Και είπατε και πάλι ότι το υπογραμμίσατε αυτό αναφερόμενος και σε προκλήσεις και ευκαιρίες. Εγώ θα σταθώ στις προκλήσεις. Ποιες είναι οι πιο σωματικές προκλήσεις και θα ήταν θετικό το ΝΑΤΟ να έχει πιο ισχυρή παρουσία στην ε, ε, νότιο-κινέζικη θάλασσα. Δεύτερον, κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ο ρόλος ε, του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά όλο αυτό το χαμό που έχουμε στη Λιβύη. Και τρίτον, υπάρχει αυτή η έννοια που είναι της μοδός, στρατηγική αυτονομία. Την ανέφερε ο κύριος Γκάλερ. Κάποιες φορές συνήθως υπάρχει μια αντινατοική χρειά σε όλη αυτή την έννοια. Ποιος είναι ο δικός σας αγαπημένος ορισμός της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαριστούμε. Ζερόμ Βιβιέρ από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Μια στιγμή περιμένετε να βάλετε ακουστικά του Γενικό Γραμματέας. Ε, Καλημέρα, έλεγα λοιπόν ότι πολλά μπορεί να πει κανεί για τον ΝΑΤΟ και για τη λήξη του ψυχρού πολέμου. Σα άκουσα και είχα την εντύπωση ότι άκουγα έναν εκπρόσωπο των ΗΠΑ, αλλά εντάξει δεν πρέπει να μα εκπλήσει γιατί η Αμερική είναι αυτή που συνεισφέρει περισσότερο και εσεί ε, βέβαια προστατεύετε τον προπολογισμό σα. Όμω τα πρόσφατα ε, που είπατε για την Τουρκία είναι αυτό που βάζει πρόβλημα. Η Τουρκία είναι ένας ενεργός ε, πρωταγωνιστής στην κρίση της Συρίας και της Λιβύης και υπάρχει ο κανόνας της ελληνικής. Οπότε τι θα γίνει με τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει θέμα κυριαρχίας της Κύπρου. Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Ερντογκάν ανοιχτά ανακατεύεται στα αισθήματα της Γαλλίας και της Γερμανίας μέσω των τουρκικών κοινοτήτων εκεί. Ε, χρησιμοποιεί τους μεταναστάτες για να απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγκάζεται τελικά να πληρώνει. Αυτή είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι δεν έχει νόημα αυτή η συμμαχία, οπότε θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η δικιά σας στρατηγική. Ε, επαναλαμβάνω, δεν βλέπω να καλύπτονται τα συμφέροντα της Γαλλίας εκεί. Ευχαριστούμε. Έχουμε δύο συντονιστές από τη ECR. Μήπως να δώσω το λόγο στο Τζέφρι Φανόρντεν, ε, κυρία Φωτίγκα, και όχι σε εσά. Και δεν ξέρω, ίσως είναι η τελευταία φορά που έχει την ευκαιρία να πάρει το λόγο ως μέλος της ε, ΑΦΕΤ. Ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε και δύο, λέει κυρία Φωτίγκα. Αλλά ναι, ας πάρει εκείνο πρώτα το λόγο. Ωραία, καλές ε, σχέσεις με την άλλη πλευρά της μάχης. Κύριε Φανόρντεν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα, εδώ είμαι. Καλώς ήρθατε ήμουνα εγώ ε, υπουργό στο ΝΑΤΟ, οπότε ε, ναι, σας καλωσορίζω θερμά εδώ. Δύο θέματα θέλω να θίξω, τα οποία έχουν ε, ήδη θίξει οι συνάδελφοι, αλλά ίσως η δικιά μου προσέγγιση να είναι ελαφρά διαφορετική. Φοβούμαι ότι υπάρχουν δύο εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή θα μπορούσαν να απειλήσουν την ενότητα στη συμμαχία. Το πρώτο είναι η προσπάθεια για στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια αποκλειστική προσέγγιση που έχει να κάνει με την άμυνα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε αυτό να διχάσει ε, τους Ευρωπαίους από την υπηρετική Ευρώπη και τους Αμερικανούς συμμάχους μας από την άλλη. Το άλλο είναι το ότι δεν μας απασχολούν τα συμφέροντα της Τουρκίας και η ψυχρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ίσως οδηγήσει την Τουρκία να ψάξει συμμάχους αλλού. Την Τουρκία πρέπει να την κρατήσουμε στο πλευρό μας και εμένα με ανησυχεί αυτή η τάση που αναγνωρίζω. Θα ήθελα πολύ τα σχόλιά σας από αυτού. Ευχαριστούμε Τζέφρι. Από την ΚΟΕ, αν δεν θέλει κανείς... Α, παρακαλώ, την ΚΟΕ. Ένας από τους δύο. Καλά, οι κυρίες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα Στόλτεμπερκ. Εσείς αναφερθήκατε ε, σε αύξηση των επενδύσεων όλων των χωρών ε, προς τον ΝΑΤΟ και ότι αυτό είναι θετικό. Εγώ αμφιβάλλω κατά πόσο είναι θετικό να βάζουμε όλο και περισσότερα χρήματα στην άμυνα και στον εξοπλισμό. Αναφερθήκαμε στους Αμερικανούς στρατιώτες στη Πολωνία και σε διάφορες χώρες. Και όταν μιλάτε για επίση όρε εταιρική σχέση, ποιοι είναι αυτοί οι εταίροι που είναι επίση όρε. Θα ήθελα να μας δώσετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Δεύτερον, η σύνδεση με την ΠΕΣΚΟ θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να το κάνουμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ξοδεύουν 340 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς είμαστε τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ όμως. Και πριν από την τελευταία διάσκεψη του ΝΑΤΟ, ο πρόεδρος Μακρόν αναφέρθηκε σε εγκεφαλική νέκρωση. Οπότε καταλαβαίνετε πώς συμπεριφέρονται πια οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λοιπόν πόσο εκτιμάτε το μέλλον του ΝΑΤΟ. Κύριε Γενική Γραμματέα, πρώτος γύρος. Εγώ αισθάνθηκα λίγο σαν την ακρόση του κύριου Μπορέλ. Ε, δεν ξέρω, εκείνος ίσως είχε λιγότερη πίεση από αυτή που έχετε εσείς για να απαντήσετε. Ας αρχίσουμε με την ερώτηση του Κρίς Πέτερ και θα καταλήξουμε στα σχόλια της κυρίας Δεμιρέλ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αν μη τι άλλο να θίξω όλα τα θέματα που θίξατε κι εσείς. Πρώτον, ο κύριος Πέτερς με ρώτησε για τα σχόλια του κύριου Τραμπ που μίλησε για περισσότερο ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή. Τι εννοεί. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Εδώ συζητάμε. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία μέσα στο ΝΑΤΟ αλλά και με τους εταίρους μας και με τους εταίρους μας στην περιοχή Ιράκ, Ιορδανία κλπ. για το κατά πόσο αν το ΝΑΤΟ κάνει κάτι περισσότερο, τι θα ήταν αυτό. Οπότε δεν είμαι σε θέση να σας δώσω συμπεράσματα, απλώς να σας περιγράψω τη διαδικασία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να κάνει περισσότερα, αλλά όχι σε θέσεις μάχης. Δηλαδή, το θέμα που εξετάζουμε δεν είναι κατά πόσο θα ξεκινούσαμε νέες μάχες, όχι. Είναι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να αποφεύγαμε τέτοιες μάχες. Η πρόληψη είναι καλύτερη από την παρέμβαση. Αν δούμε το Ιράκ, πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν δράσουμε τώρα, θα αναγκαστούμε ίσως να ξαναμπούμε σε μάχες. Εγώ ήμουνα κατά το 2003 ως πολιτής και πολιτικός της Δανίας. Ήμουνα κατά. Η Δύση όμως μάλλον έφυγε νωρίς, γιατί μετά πήγε το ISIS. Οπότε στην Ευρώπη πρέπει να στηρίξουμε τη δράση του 2014 που ήταν για την καταπολέμηση του ISIS από την αριστερά μέχρι τη δεξιά συμφωνήσαμε όλοι ότι δεν μπορεί να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να βλέπουμε να αναπτύσσεται το ISIS, να μεγαλώνει και να σκοτώνει, να βιάζει και να απειλεί όχι μόνο ε, τον έλεγχο μιας μεγάλης επικράτειας αλλά ακόμα και της ε, ε, Βαγδάτης και παραπέρα. και κλπ υπήρξε ευρεία συμφωνία ότι έπρεπε να επανέλθουμε στα πεδία της μάχης με βομβαρδισμούς, με χερσές δυνάμεις επίσης κάποιες και πλήρωσε το ΝΑΤΟ αλλά και ε, το Ιράκ πλήρωσε μεγάλο τίμημα και οι πολίτες εκεί. Η απελευθέρωση της Ράκα χρειάστηκε σκληρές προσπάθειες και πολλοί πλήρωσαν το τίμημα αυτής της απελευθέρωσης. Και απλοί πολίτες, άμαχος πληθυσμός. Δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό, πρέπει να το αποτρέψουμε και να δημιουργήσουμε και ικανότητες επιτόπου, ώστε να μπορούν να φροντίσουν να μην επανέλθει το ISIS. Και στο Ιράκ αυτό πρέπει να κάνουμε, να καταρτήσουμε περισσότερες δυνάμεις. Δεν λέω ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα, αλλά αν δεν το κάνετε, τότε θα έχουμε σίγουρα ένα μεγάλο πρόβλημα. Και μετά μπορεί να καταλήξουμε πάλι σε συμμετοχή σε μάχες. Πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να αποφύγουμε κάτι τέτοιο στο Ιράκ ε, και αλλού. Πρέπει να χτίσουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε ικανότητες επιτόπου, να καταρτήσουμε δυνάμεις εκεί. Το ΝΑΤΟ μπορεί να το κάνει και μπορεί να το κάνει και περισσότερο και θα έπρεπε να το κάνει περισσότερο. Έχουμε μια συμμαχία που προσφέρει τέτοια κατάρτιση και οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούμε να το κάνουμε μαζί. Το συζήτησα με τον Πρωθυπουργό του Ιράκ την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Πρόεδρο αυτή τη εβδομάδα. Περιμένουμε πρόσκληση από το Ιράκ. Αλλά μας το ζητάνε. Μας το ζητάνε. Γιατί καταλαβαίνουν και εκείνοι ότι χρειάζεται πιο ισχυρή ε, δύναμη επιτόπου για να μην επιστρέψει ο ISIS. Οπότε η απάντησή μου είναι, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να σας δώσω μια ακριβή απάντηση, γιατί είμαστε στη διαδικασία, αλλά αυτό που εξετάζουμε είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί και κυρίως στο Ιράκ για να ενισχύσουμε τις τοπικές ε, δυνάμεις. Απάντησα και σε άλλους που με ρωτήσανε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Έπειτα με ρωτήσατε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα αποφασίσω εγώ. Εγώ είμαι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Δεν θα αρχίσω εγώ να υπαγορεύω αν ε, το έκανα ακόμα και στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, ε, θα είχα μεγάλο πρόβλημα. Δεν το κάνω λοιπόν, οπότε δεν θα το κάνω και εδώ. Έπειτα, πολλές ερωτήσεις προσπαθώ να τις ε, ομαδοποιήσω για τη στρατηγική αυτονομία. Εγώ στηρίζω περισσότερες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμυνά της. Και γιατί όχι. Το ΝΑΤΟ ζήτησε περισσότερες προσπάθειες και το κάνει εδώ και χρόνια αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίσει να επενδύει σε περισσότερες και νέες ικανότητες, να πανέ περισσότερα για την άμυνα, να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, τόσο το καλύτερο. Αυτό θέλουμε, κανένα πρόβλημα. Συγχρόνως όμως, λέω και η κυρία Φοντερ Λάιεν τα είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι εδώ. Δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κάτι εναλλακτικό ε, με το ΝΑΤΟ. Όχι. 90% και παραπάνω του κόσμου που ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από χώρες ΝΑΤΟ. Οπότε η Ευρωπαϊκή Άμυνα ε, προφανώς έχει να κάνει και με το ΝΑΤΟ. Και είναι θετικό να υπάρχει. Εφόσον, όπως είπα, δεν υπονομεύει το ΝΑΤΟ ούτε επικαλύπτει τα όσα κάνει το ΝΑΤΟ, αλλά το συμπληρώνει. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περιθώριο για κάτι τέτοιο, βεβαίως. Για να βοηθηθούν οι δράσεις του ΝΑΤΟ, βεβαίως. Αν όμως αυτά τα νέα συστήματα δημιουργήσουν νέους φραγμούς και εμπόδια στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τότε όχι, θα ήταν επικίνδυνο. Αναφέρεται εξάλλου στις συνθήκες ότι για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ε, άμυνα. Είναι θέμα μεγέθους, όπως καταλαβαίνετε. 80% των ε, χρημάτων τώρα που θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο θα έρχονται από εκτός χώρες. Ηνωμένε Πολιτείε, Καναδά και παίζει ρόλο η γεωγραφία. Γιατί αν κοιτάξετε στο βορρά, στο βορρά είναι σημαντικές για, την ε, βόρεια, για το βόρειο Ατλαντικό, παρόλο που υπάρχουν πολλοί πάγοι εκεί. Η Τουρκία είναι στρατηγικά πολύ σημαντική χώρα ε, στον νότο για το ΝΑΤΟ. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσφέρει συλλογική άμυνα για την Ευρώπη. Πρέπει από κοινού να γίνεται η προσπάθεια αυτή από ολόκληρη την Ευρώπη με την ε, Βόρειο Ατλαντική Συμμαχία. Το θέμα της στρατηγικής αυτονομίας. Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο καλύτερος ορισμός για μένα, καλά πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι δεν θα βρω εγώ τον ορισμό, αλλά η γνώμη μου είναι ότι πρόκειται για μία έννοια που δεν είναι απόλυτα σαφής. Στρατηγική όταν λέμε σκεφτόμαστε κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό. Και όταν ακούμε τη λέξη αυτονομία σκεφτόμαστε απομόνωση, μεμονωμένο κάτι. Γι' αυτό δεν είναι καλός αυτός ο ορισμός, η ονομασία αυτή. Αλλά ίσως υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να βρούμε. Αλλά, αν πάση περιπτώσει, δεν είμαι εγώ που θα το βρω αυτό, εσείς. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσης της Ευρώπης από τη Βόρεια Αμερική θα αποδυναμώσει και την Βορειοατλαντική Συμμαχία, αλλά και την Ευρώπη. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν θα δεχόντουσαν την αποδυνάμωση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οπότε αν προσπαθείτε να απομακρύσετε την Ευρώπη από, την, από το ΝΑΤΟ, ε, αποδυναμώνετε την Ευρώπη, κάνετε κακό και στην Ευρώπη. Εγώ είμαι Ευρωπαίος και πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο φορές αγωνίστηκα, απέτυχα, για να τα καταφέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα βρείτε πολλούς να κάνουν εκστρατεία υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο ένθερμα όπως εγώ. Πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι σαν κάτι εναλλακτικό ως προς την Βορειοατλαντική Συμμαχία. Τουρκία και όλα τα άλλα. Απάντησα σε έναν βαθμό, αλλά συνεχίζω. Πήγα στην Κωνσταντινούπολη δύο μέρες μετά την ε, ε, επέμβαση αυτή και μίλησα και με τους υπουργούς και με τον Ερτογάν και εξέφρασα την βαθιά μου ανησυχία και τις συνέπειες αυτής της στρατιωτικής επέμβασης. Και είπα επίσης πόσο σημαντικό είναι η αποκλιμάκωση και να σταματήσουν οι σειράξεις. Υπάρχουν συμφωνίες με την Τουρκία, παραμένουν προβλήματα, αλλά πάντως η εμπόλεμη σύραξη εκεί έχει καταπραγηθεί πολύ σημαντικά. Χρειάζεται μια πολιτική λύση, μια ειρηνική λύση. Και εγώ στηρίζω αυτές τις προσπάθειες. Και το είπα. Στο ΝΑΤΟ υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στη Βόρεια Συρία. Αυτό είναι αλήθεια. Το ΝΑΤΟ είναι μια πλατφόρμα όπου συμμετέχουν οι διάφοροι σύμμαχοι και συζητούν και προσπαθούν να καταλήξουν σε κάτι και όταν διαφωνούν. Το καλό είναι ότι συμφωνούμε σε πολλά σημαντικά θέματα όσον αφορά την Συρία. Το θέμα της στήριξης στο Ιράκ, και ότι όλοι συμμετέχουμε στο συνασπισμό για την καταπολέμηση του ISIS. Και είναι σημαντικό σύμμαχος η Τουρκία. Κανείς δεν έχει αντιμετωπίσει τόσες επιθέσεις όσες η Τουρκία από τον ISIS. αν δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το χώρο της Τουρκίας, δεν θα είχαμε πετύχει όσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στην καταπολέμηση του ISIS. Brexit τώρα. Δεν θα αλλάξει τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με τον ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Με ρωτάτε τι πρέπει να κάνουμε για να παραμείνουν κοντά μας. Να, άλλο ένα επιχείρημα για την στενή συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε μια χώρα είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε όχι, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι κοντά. Όλοι οι σύμμαχοι, ανεξάρτητα από το κατά πόσο συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχουν εταιρικέ σχέσεις, ναι. Ε, για τον κύριο Πετικόφερ, Κίνα. Η ιδέα δεν είναι το ΝΑΤΟ να πάει στη Νότια Κινέζικη θάλασσα, αλλά να επενδύει το ΝΑΤΟ στις υποδομές, γιατί η Κίνα ξέρουμε ότι το κάνει στην Αφρική και αλλού. Το θέμα δεν είναι εμεί να εξαπλώσουμε τον ΝΑΤΟ, αλλά ότι η Κίνα φτιάχνει συστήματα ε, με τα οποία μπορεί να πλήξει όλες τις ε, χώρες του ΝΑΤΟ. Λιβύη. Είμαι υπέρ της στήριξης των προσπαθειών για λύση. Χαίρομαι για τη διάσκεψη στο Βερολίνο. Χρειάζεται κατάπαυση ε, πυρός και χειρία και όχι όπλα στη Λιβύη. Αυτή είναι μια σύντομη απάντηση για το πώς να αντιμετωπιστεί η δύσκολη κατάσταση στη Λιβύη. Χρειάζεται πολιτική λύση να διαπραγματευτούμε. Το θέμα της Λιβύης δείχνει, για καλό ή για κακό, το θέμα της συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ. Όταν ξεκίνησε η επιχείρηση για τη Λιβύη, ξεκίνησε, για τη ξεκίνησε χωρίς τον ΝΑΤΟ. Εγώ στο Παρίσι και θυμάμαι ότι ήμουνα με τον Δανό Πρωθυπουργό, με τον Κάμερον, και ήταν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν λέω ότι ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά μετά από λίγο αντιληφθήκαμε ως Ευρωπαίοι ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς την βοήθεια του ΝΑΤΟ. Και μετά πήγαν οι Ευρωπαίοι στο ΝΑΤΟ και ζήτησαν βοήθεια. Ξεκίνησε η εκστρατεία από την Ευρώπη, η πρωτοβουλία ήταν της Ευρώπης χωρίς το ΝΑΤΟ, αλλά μετά από μερικές μέρες καταλάβαμε ότι δεν είχαμε την ικανότητα και ζητήσαμε βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Ηνωμένε Πολιτείε κλπ. Οπότε είτε κάποιο συμφωνεί δεν συμφωνεί με την εκστρατεία τη Λιβύης, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Το θέμα μας είναι ότι όταν χρειάζεται η Ευρώπη μπορεί να ζητήσει βοήθεια από τον ΝΑΤΟ. Όπως έγινε τότε στη Λιβύη με πρωτοβουλία όμως που είχε αναλάβει η Ευρώπη. Στη συνέχεια, ε, έχω απαντήσει στο επόμενο. Τι άλλο, Τουρκία είπα. για τον Defender 2020. Είναι μια σημαντική άσκηση διότι θα δείξει την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξει και να προστατεύσει την Ευρώπη εφόσον χρειάζεται. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε το ΝΑΤΟ και ο λόγος για τον οποίο έχουμε τις εγγύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας για όλους και όλοι για έναν, είναι ακριβώς η προστασία της ειρήνης ο λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ δεν είναι να κάνει πόλεμο, είναι να αποφεύγει τον πόλεμο. Να αποφεύγει τις σειράξεις. Η ιδέα του ΝΑΤΟ είναι ότι κανονικά δεν θα πρέπει ποτέ να αναγκαζόμαστε να φτάσουμε στον πόλεμο. Θα πρέπει να τον αποφεύγουμε, να τον προλαμβάνουμε, προσφέροντας προστασία. Και αν υπάρχει κάποια επίθεση κατά μέλους του ΝΑΤΟ, θα υπάρχει ε, από την άλλη μεριά ε, βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, να δείχνουμε ότι είμαστε σε θέση να φέρουμε στρατεύματα από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι δυνατόν υπάρξει επίθεση ε, σε μέλος που βρίσκεται στην Ευρώπη χωρίς να έρθει βοήθεια από το ΝΑΤΟ. Είμαστε και δύναμη αποτροπής και άμυνα. Τον κύριο Φανόρντεν απάντησα για τη στρατηγική αυτονομία. Οι δαπάνε. ναι. Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό, προσαρμόζεται από το τέλος του ψυχρού πολέμου συνέχεια. Δεν συμφωνούμε πάντα όλοι, αλλά παρά τις διαφορές μας μπορούμε να καταλήγουμε σε αποφάσεις και να εφαρμόζουμε μέτρα για να προσαρμοζόμαστε μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για στρατιωτικές προσπάθειες, αλλά και για μη στρατιωτικές. Διάλογο, έλεγχος όπλων και αποφυγή κλιμάκωσης στη Μεσανατολή. Τώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν που πολλέ φορέ είναι σκε... πολύ σκεπτικοί για να ξοδέψουν περισσότερο για την άμυνα. Προτιμούν να πληρώσουν ε, για την υγεία, για την εκπαίδευση, για υποδομέ και όχι για την άμυνα. Και εγώ ήμουν πολιτικό, πολλά χρόνια και πάντα ήταν δύσκολο να πετύχουμε χρήματα για την άμυνα. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90 που ήμουν υπουργό οικονομικών και είχα μειώσει τον προπολογισμό για την άμυνα. Ναι, το έκανα. είναι προφανώ το δεκαετία του 90 όταν εγώ ήμουν υπουργό οικονομικών μετά τον ψυχρό πόλεμο μειώσαμε τις αμυντικές δαπάνες γιατί οι εντάσει είχαν μειωθεί. Αν όμως μειώσουμε τις δαπάνες όταν οι εντάσει πέφτουν, αντίθετα όταν οι εντάσει ανεβαίνουν θα πρέπει να αυξάνουμε και τον προπολογισμό άμυνας. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα, τότε πρέπει να δαπανίσει και περισσότερα. Το βλέπουμε, τη Ρωσία, τις παραβιάσεις που κάνει με τις, τους δικούς της πυράβλους και τις ικανότητές της. Γι' αυτό θα πρέπει να μην υπάρχει καθόλου καμία παρεξήγηση. Να μην νομίζουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να στηρίξει και να καλύψει τους συμμάχους του. Όσο το ΝΑΤΟ είναι εντάξει, κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να παραμείνει αξιόπιστη η δύναμη αποτροπής μας. Και άρα χρειάζονται περισσότερες δαπάνες για την άμυνα. Ξέρω, δεν ήμουν σύντομο, αλλά είχατε τόσο πολλέ ερωτήσεις. Θα ήθελα απευθεία να δώσω το λόγο στην κυρία Λουαζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα. Θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι σύντομη για να κλείσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων ε, που είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Δύο στοιχεία συγκρατώ που θεωρώ πολύ σημαντικά. Πρώτον, η πεποίθηση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να κάνει ε, ε, οικονομία σε ό,τι αφορά την στρατηγική του Υπάρχουν πολλές ε, απειλές και ποικίλε. Υπάρχουν ε, τρομοκρατικές προκλήσεις από την ε, Μέση Ανατολή και το Σαχέλ. Θα πρέπει να παραμείνει λοιπόν ισχυρή η προτεραιότητα, η σταθερότητα και η ειρήνη στην Ευρώπη. Αναφέρθηκαν πολλοί στην Τουρκία και την άνοδο των πιέσεων και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή που είναι κάτι ιδιαίτερα το ανησυχητικό. κρατάμε κατά νου ότι δεν έχει ε, δεν έχουμε πετύχει ακόμα τον στόχο μας πλήρως. Λοιπόν, απαιτείται περαιτέρω διάλογος. Διατηρώ επίσης ε, την απαραίτητη ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, ε, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για, την, για το συνασπισμό, τη συμμαχία και για το ΝΑΤΟ. Ε, βέβαια, στο συνασπισμό αυτών δεν έχουμε αρκετά βαρύνουσα σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εξοπλισμών. Εμείς προτιμούμε να είμαστε βέβαια στο τραπέζι διαπραγματεύσεων από ότι όχι. Το ΝΑΤΟ βέβαια δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν γυρνάμε την πλάτη στο ΝΑΤΟ φυσικά. Εμείς αναλαμβάνουμε τις δικές μας ευθύνες στην άμυνα της επίρου μας. Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε βέβαια σήμερα το ζήτημα αυτό, γι' αυτό και επενθυμίζω ότι η Υποεπιτροπή Άμυνα και Ασφάλεια θα συνεχίσει τακτικά τι ε, ανταλλαγέ απόψεων με το ΝΑΤΟ. 23 Ιανουαρίου είναι η επόμενη για τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Συμμαχία ε, και με παρουσία της Καμίγκ Grand.